Άρχεται η συνεδρίαση η οποία διακόπηκε στις 5 ε, Ιουλίου. Τα πρακτικά της συνεδρίασης της 5ης Ιουλίου έχουν μοιραστεί. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Όχι. Οπότε τα πρακτικά εγκρίνονται. Αγαπητοί συνάδελφοι, Χαίρομαι που μπορώ να σας καλωσορίσω στην πρώτη μας συνεδρίαση μετά τις ε, καλοκαιρινές ε, διακοπές. Ελπίζω να ξεκουραστήκατε γιατί οι επόμενοι μήνες οπωσδήποτε θα αποδειχτούν δύσκολοι. Ξέρετε πως ε, Τετάρτη το πρωί θα έρθει εδώ πέρα ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Μπαρόσο, για να μας μιλήσει για την κατάσταση της Ένωσης, για την άποψή του, για την κατάσταση δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως θα έχουν μια έντονη συζήτηση. Ελπίζω λοιπόν πως θα έρθετε πολύ σε αυτή την συζήτηση για να έχετε την ευκαιρία να εκθέσετε τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των ομάδων του. Πρέπει επίσης με την επανάληψη των εργασιών μας να σας μεταφέρω ορισμένες θλιβερές ειδήσει ανακοινώσεις ε,